Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ την προσοχή σας. Ε, την ε, Πέμπτη είσαστε πάντα κάπως ε, ανήσυχοι όταν δεν ξεκινάμε στην ώρα μας. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα να ξεκινήσουμε ακριβώς την ώρα μας. Mr. Carter. Yeah. Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, Αγαπητοί συνάδελφοι, βλέπω μία, ένα αίτημα για δικαστικό να μας πείτε σε ποιο άρθρο αναφέρεστε. Um, thank you, Chair. I'm... Ευχαριστώ Πρόεδρε και βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 3 θέλω να θέσω ένα δεδευτικό ζήτημα. Είναι σαφέ ε, από την παρέμβαση της κυρίας Τσάκη Φώστερ Χθε, ο κύριος Κόρμπετ ε, εκπροσώπησε με λάθος τρόπο σε ό,τι αφορά τον ρόλο του κυρίου Φερχόφστατ, ε, σε ό,τι αφορά την Επιτροπή για την διαπραγμάτευση του Brexit και πρόκειται για σοβαρό ζήτημα σε ό,τι αφορά και κλείνει δυστυχώ το μικρόφωνο του ομιλητή. Η Πρόεδρος, αγαπητέ συνάδελφε, δεν πρόκειται να ξανανοίξουμε τη συζήτηση τη χθεσινή. Και έχω άλλο ένα διαδικαστικό αίτημα από τον κύριο Βόλφ. Έχετε το λόγο. Κύριε Βόλφ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Βάσει του άρθρου 184 και του 198 άρθρου, ζητώ ως πρόεδρος να εξετάζεται το Κοινοβούλιο να δημιουργήσει μια επιτροπή για να εξετάσει την ε, χαόδη και φρικτή συμπεριφορά τη κυβέρνηση τη Σαουδική Αραβία αντί τη Ιεμένη και θα πρέπει να εξεταστούν οι σχέσει με τη Σαουδική Αραβία. Όπω γνωρίζετε, η κρίση η οποία λαμβάνει η χώρα στην Ιεμένη σήμερα φτάνει και πλήττει ένα εκατομμύριο ανθρώπου. Εκατοντάδες ανθρώποι είχαν τη ζωή τους κάθε μέρα και η Σαουδική Αραβία αποφάσισε να κλείσει τα λιμάνια, τους αερολιμένες και οποιαδήποτε άλλη με, ε, ε, είσοδο. Και δεν επιτρέπει στον κόσμο αυτό να ε, φροντίσει τα παιδιά αυτά. Υπάρχει λοιπόν ευθύνη από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό βάσει του άρθρου 198. Παρακαλώ, περάστε στο διαδικαστικό σας αίτημα, λέει η Πρόεδρος. Όχι, δεν το κάνετε. Ο κ. Παπαδημούλης έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χθες μία φωνική πλημμύρα στη χώρα μου την Ελλάδα, στα προάστια δυτικά της Αθήνας, προκάλεσε μια τεράστια φυσική καταστροφή και ήδη θρηνούμε 15 νεκρούς. Θεωρώντας δεδομένη την έκφραση της αλληλεγγύης του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και όλης της ευρωπαϊκής ένωσης προς τον ελληνικό λαό που πλήττεται από αυτή την καταστροφή και ως έκφραση συλληπιτηρίων στις οικογένειες των νεκρών προτείνω κυρία πρόεδρε να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή. Σας ευχαριστώ. Και σήμερα δυστυχώς δεν μπορούμε να τηρήσουμε ενό λεπτού γη, αλλά αυτό που είναι σαφές είναι ότι όλοι στεκόμαστε δίπλα στα θύματα των καταστροφών, μεγάλες καταστροφές και μεγάλες οι απώλειες όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ που α, αναφέρετε τα θύματα και πάντα να σας πω σας ευχαριστώ που αναφέρετε τις μειονότητες και φροντίζουμε να υπερασπιζόμαστε τις μειονότητες. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για μας. Σας ευχαριστώ που μας το επισημάνατε και που μας ενημερώσατε. Αλλά αν μου επιτρέπετε θα ήθελα τώρα να περάσω στην ενημερήσια διάταξη. Ο Πρόεδρος ε, και άλλα διαδικαστικά αιτήματα, κύριε Σλένιν. Πρόεδρε, θα ήθελα να ενημερώσω την Ολομέλεια ότι στην Τρίτη το απόγευμα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το κράτος δικαίου στη Μάλτα, μετά την παρέμβαση του συναδέλφου Γκίγκαλτ, η μετάδοση live stream στη Μάλτα διακόπηκε και κατά τη διάρκεια της ομιλίας του κυρίου Κάζα. Συνολικά 28 συνάδελφοι μίλησαν και δεν αναμεταδόθηκαν. Αυτό θεωρώ ότι αποτελεί σκάνδαλο άμευ προηγουμένου και πραγματικά παρακαλώ το Προεδρείο να ερευνήσει τις αιτίες της διακοπής της αναμετάδοσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, λέει η Πρόεδρος. Τώρα δεν βλέπουν να υπάρχουν άλλα διαδικαστικά ζητήματα και ως εκ τούτου θα περάσουμε στις εργασίες μας. Ο πρόεδρος έλαβε έτοιμα από την GUE NGL. Ο κ. Μαρτάν Σιρντεβαν ε, διορίζεται στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Αποφάσεων. Ε, παρατηρήσεις παρακαλώ, ενστάσεις. Όχι. Εγκρίνεται ο διορισμός. Και περνάμε τώρα στις ψηφοφορίες. Στις ψηφοφορίες περνάμε λοιπόν καταρχάς για ένα κοινό ψηφίσμα ε, κατόπιν ετήματος πέντε ομάδων για την ελευθερία ε, έκφρασης στη Σουδάν. Επτά